δύο εκθέσεις. Η πρώτη είναι του κυρίου Ότμας Κάρας. Πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την αύξηση της πολυμορφίας της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την έκθεση Καπανάους και πώς να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δυναμικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασία. Καταρχήν θα δώσω το λόγο στον κύριο Κάρα, στον πρώτο εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Συζητούμε τώρα την έκθεση αυτή για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, στο πλαίσιο μιας ένωσης κεφάλαια αγορών. Συνηγορώ υπέρ της ειδική στόχευσης και προσανατολισμού της ε, Ένωσης Κεφαλαιαγορών που σχεδιάζουμε. Θα πρέπει να μπορούν να δανειοδοτούνται εύκολα οι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε τίποτα λιγότερο από το οι ε, αγορές να είναι στην υπηρεσία της πραγματικής οικονομίας στην Ένωση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς επίσης και οικογενειακές είναι η ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό εδώ και καιρό είναι πάγιο έτοιμά μας και είναι ε, στην πολιτική ατζέντα η χρηματοδότησή τους, η δανειοδότησή τους και θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτό το αίτημα και να το διευρύνουμε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι μικρομεσαίες δεν είναι καθόλου ενιαίες. Έχουν πολλές διαφορές ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο, το μέγεθος, το στάδιο της ανάπτυξης, την οικονομική τους και νομική μορφή η πρόσβαση των μικρομεσαίων στην χρηματοδότηση θα πρέπει να εξασφαλίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της εταιρείας η δανειοδότηση εδώ, οι χορηγήσει εξακολουθούν να παραμένουν σημαντική πηγή χρηματοδότηση για τι μικρομεσαίες. Γι' αυτό απαιτούμε η σημερινή διευκόλυνση για τραπεζικά δάνεια στι μικρομεσαίες επιχειρήσει να παραταθεί και να διευρυνθεί. Προσωπικά, στον κανονισμό για τις τράπεζες το 2013 φρόντισα η δυνατότητα αυτή για πιο ευνοϊκές ε, προϋποθέσεις για τις μικρομεσαίες να θεσπιστεί καν. Και θέλουμε αυτός ο υποστηρικτικός παράγων, επαναλαμβάνω, να παραταθεί και να επεκταθεί. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν φταίνε για την κρίση, ούτε είναι υπέτη. Οπότε θα πρέπει ε, αυτό το supporting factor, ο υποστηρικτικός παράγων, να ε, παραταθεί. Και είναι και θέμα δικαιοσύνης, είναι και θέμα κοινή λογικής, για να μπορέσουμε να δώσουμε όθηση στην οικονομία η έκθεση είναι 41 σελίδες. Ένα τρίτο ε, έχει να κάνει με τη δημιουργία ε, της μόνο απευθυντικής λεγόμενης θηρίδας, το one-stop shop. Σε κάποια, κάθε χώρα θα πρέπει να υπάρχει μία θηρίδα για να ενημερώνει για το πώς, ε, στήνεις, το πώς ιδρύεις μια επιχείρηση. Με απλό τρόπο σε κάθε κράτος μέλος από την αρχή να ξέρει ε, που βαδίζει μια εταιρεία και να μπορεί σε ένα ενιαίο φορέα να απευθύνεται. Το δεύτερο, ε, κεντρική τράπεζα δεδομένων όπου να καταθέτουν ε, τα σχέδιά τους, τα επιχειρηματικά και τις ανάγκες της χρηματοδοτικές οι μικρομεσαίες. Έτσι με τρόπο απλούστερο μπορεί η Ευρώπη να παραμένει σε επαφή με επενδυτές. Και τελευταίο αίτημα προκατακτικά έτσι πριν αρχίσει η συζήτηση, είναι η δημιουργία προγραμμάτων και έργων έτσι ώστε να ε, μπορούν να χρηματοδοτούνται οι νέοι επιχειρηματίες. Μόνο όποιος έχει ε, γερή οικονομική βάση τολμάει το καινούριο και αναλαμβάνει και κίνδυνο. Ε, για να υπάρχει μια μαγιά να ξεκινούν επιχειρήσεις νέοι άνθρωποι. Επαναλαμβάνω, η έκθεσή μου είναι 41 σελίδες και θέλουμε ε, η Ένωση κέφαλε Αγορών να εστιάσει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ε, να μην καούν και τα χλωρά μαζί με τα ξερά. Η δανειοδότηση, η τραπεζική να παραμείνει με τις διευκολύνσεις και με απλοποίηση για να μπορούν οι ε, νέοι μας να ιδρύουν επιχειρήσεις. Παρακαλώ να υποστηρίξετε την έκθεση. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη κύριε Κάρας. Και τώρα ο έτερος των συγητών, ο κύριος Κρασνοντεύσκη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για την βοήθεια που μου έδωσαν στην προετοιμασία αυτής της έκθεσης. Είχαμε κοινού στόχους και είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα θέμα μεγάλης σημασίας. Η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ευρωπαϊκή οικονομία είναι προφανής. Το 90% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι μικρές ή μεσαίες. Δημιουργούν σε μεγάλο βαθμό στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Το 2014, 71% των ε, θέσεων απασχόλησης στον ε, μη χρηματοπιστωτικό τομέα προερχόταν από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η πρωτοβουλία αυτή να στηρίξουμε την ανάπτυξη τους και να στηρίξουμε την αγορά αυτά στην οποία ενεργοποιούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σήμερα βλέπουμε ότι οι δυσκολίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, για να έχουν πρόσβαση στα εργαλεία των ε, κεφαλαγορών είναι σημαντικές. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ε, θέσεις εργασίας, βρίσκονται όμως σε πολύ άνηση θέση σε πολύ δύσκολη θέση σε σχέση με τις μεγάλες πολυεθνικές ε, εταιρείες και τους μεγάλους ομίλους. Η θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα κράτη-μέλη βεβαίως είναι το αντικείμενο αυτής της έκθεσης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι θύματα ρυθμίσεων που διαρκώς αλλάζουν κάποιων ε, αποφάσεων δικαστικών ε, άδικων και σκληρών και διαδικασιών διοικητικών που περιπλέκουν εξαιρετικά την ε, καθημερινή τους εργασία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές συνέπειες όλων αυτών επί των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπάρχουν πολλές διακρίσεις κατά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν πολύ ισχυρότερη θέση και συγκριτικά πλεονεκτήματα. αντιμετωπίζουν σημαντικό γραφειοκρατικό άχθος, πολλές ε, ρυθμίσεις και βεβαίως αντιμετωπίζουν και το θέμα του κόστους σε σχέση με τις ε, μεγάλες πολυεθνικές περιορισμένο προσωπικό που δεν τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις ε, διοικητικέ ε, διαδικασίες με τον ίδιο τρόπο. Πολλές φορές τους ε, λείπουν μάλιστα και τα επαγγελματικά προσόντα και οι δεξιότητες. Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε και τα ειδικά προβλήματα της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης με τις μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους αλλά και την ε, Νότια Ευρώπη, τις χώρες της Νότιας Ευρώπης με πολύ δύσκολη πρόσβαση στις ε, κεφαλαίες Πολλές περιφερειακές χώρες έχουν σημαντικά προβλήματα με την φυγή των εγκεφάλων, με τους νέους ε, πτυχιούχους οι οποίοι εγκαταλείπουν τις χώρες αυτές για να ε, βρουν δουλειά κάπου στη Βόρεια Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Σας παρακαλώ, μπορείτε να ολοκληρώσετε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντομπρόφσκης. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Βουλευτέ, η προτεραιότητα της Κομισιόν είναι ενίσχυση της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας. Αυτέ τις προσπάθειες καταβάλει. Και συζητάμε τώρα για την βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κάτι το οποίο είναι κεντρική σημασία στην ενωμένη αγορά μας. Να ευχαριστήσω τους συζητητές και όλους τους κοιοδείς για τη σφαιρική τους προσέγγιση όσον αφορά τις, προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες και τις ενδεχομένες πιθανές δράσεις. Σήμερα η Κομισιόν έβγαλε μια ανακοίνωση για την κεφαλαία αγορά. Είναι ένα σημαντικό σημείο του θεματολογίου μας για την ενίσχυση των θέσεων εργασία στην Ευρώπη. Ήδη έχουμε κάποιες δράσεις που μπορούν να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες. Εδώ έχουμε ας πούμε το καθεστώ των επιχειρήσεων και δυνατότητα άντληση κεφαλαίων από τι κεφαλαίε Θα πρέπει να έχουμε απλέ απλές και ενοποιημένες προδιαγραφές για αυτά τα θέματα. Επίσης θα πρέπει να εφαρμόσουμε σωστά και τους κανονισμούς για την ε, κοινωνική επιχειρηματικότητα και καλωσορίζουμε την υποστήριξη που δώσατε στην έκθεση του κύριου Κάρας για αυτή και για μελλοντικέ νομοθεσίε. Χρειαζόμαστε να υπάρξει πρόοδο σύντομα και είναι τώρα στιγμή ακριβώ για να εφαρμόσουμε σε αυτές τις πρωτοβουλίες μας. Θα πρέπει να επιταχύνουμε όπου υπάρχει περιθώριο στην κεφαλαία αγορά και να δώσουμε στις επιχειρήσεις την βεβαιότητα που χρειάζονται για να επενδύσουν παντού και για τα συστήματα σταξιδεώτησης και τον ενίο χαρακτήρα αυτών των κεφαλαίων αγορών. Θα πρέπει εδώ να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την καινοτομία και επίσης καλωσορίζουμε και την καθεστώτα που αφορούν το, την πτώχευση και τα σχέδια δράσης. Είχαμε ξεκινήσει φέτος και μία διαβούλευση για την δημιουργία μιας νέας αγοράς συντάξεων και αναμένεται νέα νομοθεσία από αυτού. Επίσης, η Κομισιόν σύντομα θα υποβάλει προτάσεις για την διάρθρωση των επιχειρήσεων και θα θέλαμε επίσης να είμαστε και πιο τολμηροί σε κάποιους τομείς. Να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ακριβώς για να προωθήσουμε τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Επ' αυτού θα συγκροτήσουμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ακριβώς για αυτά τα θέματα για να δούμε ακριβώς πώς θα μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά με ασφαλή τρόπο σε όλη την Ένωση. Η ανακοίνωση η σημερινή θα αυξήσει τη χρηματοδότηση για όλες τις επιχειρήσεις νομίζω περιλαμβανομένων και των μικρομεσαίων. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τη χρηματοδότηση, τη χρηματοδότησή τους υπό το Ταμείο Αυσταρικής Χρηματοδότησης και έχουμε γύρω στις 200 ε, συμφωνίες με χρηματοοικονομικούς διάμεσους που αφορούν ακριβώς αυτό το είδος επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά, ο τραπεζικός ε, δανεισμός παραμένει η κύρια μορφή χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες. Θέλουμε να υπάρχει διεύρυνση ενός ευνοϊκού οικονομικού πλαισίου χρηματοδότηση αυτές τις επιχειρήσεις και στο τωρινό οικονομικό πλαίσιο χρειαζόμαστε όσο περισσότερο από ό,τι ποτέ την ενιαία κεφαλαία αγορά. Και γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να επιταχύνουμε τη δουλειά μα. Ο κ. Κανοντζεύσκη επίση τονίζει την ανάγκη για τι μικρομεσαίες και τι startup όσον αφορά τι δομικέ μεταρρυθμίσει. Συμμεριζόμαστε βεβαίω αυτές τις ανάγκης μεταρρύθμιση στις δεξιότητε που θα πρέπει να συνοδεύουν και τι μικρομεσαίες και η υποστήριξη των καινοτόμων startups είναι απαραίτητο. Όμως η επιχειρηματικότητα θα πρέπει να αποτελεί μια ελκυστική μορφή επιχειρηματικότητα και για τους ε, μη ευνοημένους. Η Κομισιόν θεωρεί ότι η αυτοαπασχόληση δεν είναι πανάκια και η ποιότητα των θέσεων ε, απασχόλησης της δουλειάς που υπάρχει θα πρέπει να είναι αντικείμενο που μας απασχολεί. Θα πρέπει να ασχοληθούμε, ας πούμε, με την άτυπη εργασία και με την αδήλωτη εργασία στην Ευρώπη. Οι εκθέσεις αναφέρονται και σε άλλους ε, τομείς στα πλαίσια των ευρωπαϊκών πυλώνων όπου εδώ και πάλι για τις μικρομεσαίες θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Κυρία Πρόεδρε και κύριοι βουλευτές, είμαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ε, σχόλιο και για παραγωγική δουλειά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Πριν αρχίσει η συζήτηση, θα ακούσουμε τους ομιλητές ε, που γνωμοδοτούν εξ ονόματος των Επιτροπών. Από την Επιτροπή Προεπολογισμών, ο κύριος ε, Κούσμιουκ, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, λαμβάνω το λόγο για να επικεντρωθώ στα εξή σημεία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Ε, παράγουν πάνω από 50% του ΑΕΠ στην Ένωση και απασχολούν το 70% του εργατικού δυναμικού. Έχουν μεγάλες διαφορές. Υπάρχουν πολύ μικρές επιχειρήσεις, μεγαλύτερες και μεσαίες, με διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα. Επίσης, η πιο σημαντική πηγή χρηματοδότησής τους είναι και παραμένει η τραπεζική ε, δανειοδότηση. Και εκεί έχουμε διαφορές ανάλογα με το είδος της εταιρεία και το είδος της χρηματοδότησης, της χορήγησης από την τράπεζα. Πολλές μικρομεσαίες ε, χρηματοδοτούνται και από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κόσμε αλλά και από τις χρηματαγορές. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, δώσει ε, ε, πάρα πολλά χρήματα στην Πολωνία για αυτό το σκοπό. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Επόμενη Επιτροπή. Δεν βλέπω τον κύριο Ζουλό, δεν θα ακούσουμε την Περιφερειακή Επιτροπή λοιπόν. Οπότε θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μοργάνο που θα μιλήσει εξ ονόματος της Επιτροπής ε, Πολιτισμού. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Υπόθηκε ότι οι μικρομεσαίες είναι η κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Μεταξύ αυτών, οι μικροεπιχειρήσεις στον τομέα της ψυχολογίας και του πολιτισμού έχουν ένα σημαντικό ρόλο για την διατήρηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας Ευρώπης. Εκπροσωπούν το 4,5% της ευρωπαϊκής οικονομίας και προσφέρουν εργασία σε 4,5 εκατομμύρια πολιτών συγκρίσιμο με τον τομέα των ασφαλίσεων και των τραπεζών. Κυρίως έχουμε να κάνουμε με νέους μεταξύ 15-29 ετών. Χαρή επίση στην πολύ στενή σχέση είναι δύσκολο που έχουμε τις, ε, με, τα, με τα διάφορα μέρη στα οποία βρισκόνται είναι δύσκολο να μετακινηθούν. Η πρόσβαση λοιπόν στην δανειοδότηση για αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ιδιαίτερα προβληματική. Πρέπει λοιπόν σε αυτή τη ε, φάση της ψηφιακής μεταξέλιξης να διασφαλίσουμε ικανότητες και την εξέλιξη αυτών των επιχειρήσεων και την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα ώστε να χρηματοδοτούνται ανάλογα με τι δυνατότητε που έχουν όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και τι δυνατότητε εξέλιξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Νίρη Άνταξ, ονόματος Επιτροπής Προϋπολογισμών και πάλι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Υπάρχουν και καλά σημεία στην έκθεση αυτή, αλλά είναι απογοητευτικό ε, που δεν κάνει καθόλου κουβέντα για τις διαφορετικές ανάγκες που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως γνωρίζουμε, ε, επλήγησαν ε, σφοδρά από την κρίση. Από το 2008 έχουν μειωθεί οι υπηρεσίες προς μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις. Δεν είναι δίκαιο αυτό ε, να επιβαρύνονται μικρομεσαίες ενώ οι κολοσσοί ε, οι πολυεθνικές κάνουν συμφωνίες με την ελλαδική κυβέρνηση. Προφανώς εννοώ την υπόθεση της Apple. Η Ένωση Κεφαλαίου Αγορών βέβαια δεν είναι η απάντηση ε, οι δημόσιες τράπεζες, τα χαμηλότοκα ή τα άτοκα δάνεια είναι πολύ συγκεκριμένα μέτρα και πολύ σημαντικά για να αναπτυχθεί αυτός ο ευαίσθητος και έφραυστος τομέας. Δεν θα πρέπει να είναι εμπόδιο η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος της οικονομίας, προωθούν την τοπική ανάπτυξη και δημιουργούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα... Ψάχνω τον κύριο Νόβακοφ, αλλά δεν τον βλέπω ούτε εκείνον. Μάλλον κουραστήκαμε. Λοιπόν, εδώ τελειώνουν οι γνωμοδοτήσεις των επιτροπών και ακολουθούν οι ομιλητέ εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Κλούν, εξ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Κνάστοντεύσκη, τον ε, εισηγητή μας, για την έκθεσή του και για την υπομονή που έδειξε απέναντι στους κοιόδης εισηγητές για να καταλήξουμε σε μια απάντηση συνεκτική και συνεπή για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως είπε και ο ίδιος, θα πρέπει να επικεντρωθούμε πάρα πολύ σε αυτές τις εταιρείες και ιδιαίτερα στις νεοφυείς, στις startups θα πρέπει να υποστηριχθούν από την αρχή, γιατί ε, ε, είναι σημαντική η πρώτη φάση της ζωής τους, η πρώτη και η δεύτερη χρονιά. Ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι οι μικρομεσαίες για την οικονομία μας, ε, πόσα εκατομμύρια εργαζομένους έχουν στην Ευρώπη. Σήμερα σε προηγούμενες συζητήσεις μιλήσαμε πολύ για τις πολυεθνικές. Θα πρέπει να πούμε ότι οι πολυεθνικές οι ίδιες υποστηρίζουν ε, την ίδρυση μικρομεσαίων γιατί πολλές μικρομεσαίες εξαρτώνται από την ύπαρξη των πολυεθνικών γιατί είναι προμηθευτές, υπεργολάβοι, ε, τους ε, προμηθεύουν εξαρτήματα, ανταλλακτικά και υπηρεσίες και άλλα. Έχουν πολύ σημαντικό ρόλο. Μείωση της γραφειοκρατίας ζητεί η ε, έκθεση και της άχρηστης γραφειοκρατίας. Δεν θέλουμε περισσότερη ρύθμιση, θέλουμε πιο ευφυή, πιο έξυπνη και όχι εξαιρέσεις. Όποιος ε, είναι στην αγορά μικρός, μεγάλος ή μεσαίος θα πρέπει να υπόκειται σε κανόνες. Δεν λέμε να μην υπάρχουν κανόνες, αλλά είναι ευφυής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας διαβεβαιώνει ότι θα μειώσει το γραφειοκρατικό άχθος και καλά θα κάνει να τηρήσει αυτές τις δεσμεύσεις Να είναι πιο εύκολο και πιο φθηνό να στείλεις μια εταιρεία, να προσλαμβάνεις κόσμο. Ακούσαμε πολλά και για το μισθολογικό κόστος και τα λοιπά. Ναι, είναι κόστος η μισθή, τι να κάνουμε, αλλά η εργασία είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο κάθε επιχείρησης, κάθε εταιρεία, ιδιαίτερα της μικρομεσαίας και δεν μπορεί να υπάρχει περικοπή εκεί στο μισθολογικό κόστος. Υπάρχει ασυμπίεστο κόστος ε, για τη ζωή των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να τους κόβουμε συνέχεια το, το μισθό. Υπάρχουν και άλλες δαπάνες, ε, νίκια κτλ. που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ο κύριος Σάιμον για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Τον κύριο Κάρα, στην την έκθεσή του και για την συνεργασία στην οποία βρίσκαμε, βρήκαμε κοινό πεδίο και συνεννόηση για τη φύση των προβλημάτων και τους τρόπους λύσης τους. Βέβαια, κάθε δεκαετία έχουμε τις ίδιες συζητήσεις για θέματα τα οποία παραμένουν. Εγώ από τα West Midlands στην Αγγλία έχουμε 378.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αριθμός ο οποίος αυξάνεται συνεχώς και παρόλα αυτά μόνο το 26%, 26 έχουν ε, αρκετούς ε, εργαζόμενους με συνεχώς μειω, μειω, μειωμένο αριθμό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε θα γίνουμε τις και να αντιμετωπίσουμε την ανεργία. Γιατί δεν κάνουν προσλήψεις όμως. Ίσως εν μέρει επειδή οι τράπεζες όσο και αν λένε ότι προσπαθούν δεν είναι αρκετά κοντά στους πελάτες τους και χρειάζεται να είναι πιο κοντά. Κυρίως όμως επειδή υπάρχει ένα κενό όπου δεν είναι εμπορικά βιώσιμο για τις τράπεζες να δανείσουν. Αυτό γίνεται. Και αυτό το κενό θα πρέπει να καλυφθεί από τον δημόσιο τομέα, από μια ευφυή προσέγγιση χρηματοδότησης. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην περιοχή μου για το πώς έχει γίνει αυτό πολύ σωστά, πολύ ωραία. Πρέπει όμως να κλιμακωθεί, να διευρυνθεί και να γίνει σε τακτική βάση. Χαζόμαστε αυτά τα one-stop shops αλλά θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε και την βάση δανεισμού, δηλαδή πέραν από τις τράπεζες να πάμε, αλλά κυρίως πρέπει να είμαστε σαφείς ότι υπάρχει ένα κενό όπου ο δανεισμός δεν είναι οικονομικής φύσης λόγω κινδύνου, αλλά λόγω κόστους και κινδύνου συναλλαγής που αφορά τις μικρομεσαίες. Αυτό λοιπόν ακριβώς το κενό θα πρέπει να καλυφθεί από το δημόσιο τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Όζοκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το 90% όλων των επιχειρήσεων και προσφέρουν τα δύο τρίτα όλων των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Η έκθεση τονίζει τη σημασία της διαφοροποίησης της χρηματοδότηση των μικρομεσαίων και υπόθηκε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξει διευκόλυνση όσον αφορά τις ε, φορολογικές και διοικητικές ε, απαιτήσεις. Ο τραπεζικός δανεισμός συνεχίζει να αποτελεί την πιο σημαντική μορφή χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με τις νόμεις ότι μπορούμε να δώσουμε στήριξη επιτυχώς και ευχαριστώ για τον εισηγηθεί για τη συνεργασία. Τώρα για την ίδια την έκθεση είμαι την, της άποψης ότι εκφράζει σωστά την τωρινή κατάσταση των μικρομεσαίων. Παρ' όλα αυτά συνεχίζω να έχω την εντύπωση ότι ένας τόσο μεγάλος ε, αριθμός ε, τροπολογιών κάνει την έκθεση πιο αδύναμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει και η Πρόεδρος. Επόμενη ομιλήτρια έχει πολύ χρόνο. Είναι η κυρία Τζεμπάλοβα. Δυόμιση λεπτά. Ναι. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κάτι που ιδιαίτερα με αφορά. Ξεκίνησα την καριέρα μου εκεί και είναι και κάτι που και σαν πολιτικό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να κοιτάξουμε τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα σας δώσω ένα κατάλογο αυτών που πρέπει κατά προτεραιότητα να γίνουν. Να υπάρξει καλύτερη προσαρμογή μεταξύ και σύνδεσμο μεταξύ αυτών που ψάχνουν ε, εργαζόμενους και των νέων πτυχίουχων. Να υπάρχουν προγράμματα όπως το πρόγραμμα Εράσμος με συνειδητοποιημένους ε, και καλά καταρτισμένους ε, νέους. Έχουμε ήδη χάσει μια ολόκληρη γενιά νέων που βρέθηκαν στην ανεργία. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί άλλη μια φορά. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξυγχρονιστούν, να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες. Να απλοποιήσουμε τους κανόνες και τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για την χρηματοδότηση και όλα τα προγράμματα Horizon 2020 ε, και τα λοιπά. Να δημιουργηθεί ένα σταθερό νομικό πλαίσιο οι υποχρεώσεις των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων να μετατραπούν σε ευκαιρίες για στήριξη και να συνειδητοποιήσουμε ότι σήμερα τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη δημιουργούνται χάρη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να στηρίξουμε την καινοτομία, την έρευνα, διότι η ανάπτυξη σε όλες τις χώρες αλλά και στην Ευρώπη στο σύνολό της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι μία από τις προτεραιότητες μου. Ευχαριστώ τους συζητητές Πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την συνεργασία στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Σέντρα Ρόντιγκες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας στην χώρα μου, στη Γαλλικία. Το 99% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες και το 96 είναι μικροεπιχειρήσεις. Έχουν λοιπόν μεγάλη σημασία. Παρ' όλα αυτά υποφέρουν από του ανταγωνισμού που προέρχεται από νεφιλελεύθερες πολιτικές που ωφελούν τις πολυεθνικές οι οποίες πληρώνουν λιγότερους φόρους. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι θέλει να λύσει τα θέματα της απασχόλησης, τότε θα πρέπει ακριβώς να υποστηρίξει τις μικρομεσαίες και να θέσει τέλος στις πολιτικές λιτότητας, τι επιχειρήσεις αυτές στο να έχουν πρόσβαση στους δημόσιους διαγωνισμού του δημοσίου και στις τράπεζες. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουμε εμπορικές συμφωνίες οι οποίες είναι αρνητικές για τις μικρομεσαίες και να αναζωογονήσουμε τομεί πρωτογενεί όπως η Αλία και η Γεωργία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να πω ο μιλήσω, κ. Κόμπορν. Κυρία Αντιπρόεδρε, ευχαριστώ. Η ενιαία, η η Ένωση Κεφαλαίου Αγορών αφορούν τις, αφορά τις, επιχει... τις επενδύσεις. Να σας πω όμως ότι οι πολιτικές ενώσεις ακριβώς αυτές θα πλήξουν τις επενδύσεις. Ο φόρος της Ιρλανδίας ήταν ένα καλό παράδειγμα γι' αυτό. Οι επιχειρήσεις, είτε μικρές είτε μεγάλες, χρειάζονται βεβαιότητα και αυτό αφορά την φορολογική τους κατάσταση. 13 δις ευρώ. Αναδρομικά άλλαξε η Ένωση με αυτό το πρόστιμο την έννοια της Κρατική ενίσχυση, όπως τη βολεύει σύμφωνα με το σχέδιό τη. Ποιο είναι το σχέδιό τη να διευκολύνει την ε, φοροδιαφυγή καταχρώντας, καταχρώνει μάλλον την δυνατότητα ελεύθερης εγκατάστασης των επιχειρήσεων. Μακροπρόθεσμα θέλουν να ακυρώσουν τους φόρους πλήρως, ώστε να μην υπάρχει κίνητρο. Τι ηρωνία λοιπόν για τον όρο επίτροπος ανταγωνισμού που αποβλέπει στην ακύρωση οποιοδήποτε ανταγωνισμού. Άσχετα με το πρόστιμο της από. Το δίδαγμα λοιπόν για το Μένο Βασίλειο ακόμα και μετά τον Brexit είναι ότι αν το Ηνωμένο Βασίλειο παραμείνει στην νέα αγορά, τότε θα υπόκειται όχι μόνο στους κανόνες των εθνικών επιδοτήσεων, αλλά και στον έλεγχο των φόρων. Η αβεβαιότητα και η φορολόγηση χωρίς εκπροσώπηση θα οδηγήσει και θα κάνει πιο αναγκαία την αποχώρηση της Βρετανίας από την αγορά. Και αυτό ακριβώς σημαίνει το Brexit. Η Ένωση είναι ξεκάθαρο δεν κατανοεί τις επιχειρήσεις, είτε είναι μικρές είτε μεγάλες είτε μεσαίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μονό, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, Πολλά ακούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λέγονται για τις μικρομεσίες. Λες και οι κλεπτοκράτες των Βρυξελών έχουν ξαναδεί μικρομεσαία. Πόσοι έχετε υπογράψει επιταγή, έχετε ψάξει για πελάτες για τις παραγγελίες. Τον κύριο Μπαρόζο τον, τον ε, προσέλαβε η Κόλμπαν Σάξ και δείχνει τη διαπλοκή και τα πλακάκια που τα έχουν κάνει οι Βρυξέλλες με τη Wall Street. 25 χρόνια υπέρ ποιου είναι ε, η αγορά για τις, των μεγάλων πολυεθνικών που δεν ευρωπαϊκές ξένα κεφάλαια έρχονται εδώ και αλωνίζουν και οργιάζουν με στρατηγικές επιχειρήσεις. Στη Γαλλία η Alstom με την General Electric, τα είδαμε, είναι επικαιρότητα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πραγματικά ε, κάνει να στενάζουν τις μικρομεσαίες. Οι μικρομεσαίες τι θέλουν, παραγγελίες. Γι' αυτό χρειάζεται εσωτερική οικονομική ζήτηση και τα κράτη να έχουν τη δυνατότητα να δίνουν δημόσια έργα στις εθνικές τους μικρομεσαίες. Και είμαστε και σκεπτικοί και επιφυλακτικοί κατά της Ένωσης Κεφαλαιογορών και την υπόθεση της χρηματοδότησης κεφαλαγορών. Είναι κυκλικές οι κεφαλαγορές, θέλουν ε, άμεση και γρήγορη ταχεία απόδοση και δίνουν λεφτά μόνο όταν πάνε καλά τα πράγματα. Εμείς που είμαστε πατριώτες θέλουμε να υποστηρίζουμε τις εταιρείε μας και σε χαλεπούς καιρούς και όχι μόνο όταν είναι ευνοϊκά τα πράγματα, να ε, περιοριστεί η κερδοσκοπία. Ε, δέχεστε μπλε κάρτα το κύριο Κόμπορν, λέει η πρόεδρος, το κύριο Μόνο, δέχεστε ερώτηση με μπλε κάρτα. Ναι. Παρακαλώ, κύριε Κόμπορν. Χωρί μικρόφωνο. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω. Ε, έχω μεγάλη συμπάθεια και συμπάσχω και με τις γαλλικές μικρομεσαίες και τα προβλήματά τους και περνάνε τα πάνδυνα. Συμφωνείτε ότι η απάντηση σε αυτό θα ήταν ε, να έρθει μαζί μας η Γαλλία και να έχουμε και το Frexit που η κυρία Λεπέν από ό,τι ακούω έχει ήδη προτείνει. Συμφωνείτε μαζί μου. Μετά το Brexit τώρα το Frexit. Ε, κύριε Μονό, ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Βλέπω ότι είστε υποστηρικτής του Brexit, προφανώς. Αυτή είναι η λύση, φυσικά. Αλλά πριν ε, τολμήσουμε ή αποπειραθούμε το Frexit, ε, το γαλλικό, θα προσπαθήσουμε παρόλα αυτά να διαπραγματευτούμε στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο για δύο-τρία κριτήρια όπως αυτά του Ηνωμένου Βασιλείου. Έξοδος από το Σέγγεν ε, και ανάκτηση της εθνικής ε, κυριαρχίας στα οικονομικά και στα νομισματικά, όπως και σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος... Ωραία. Χαίρομαι με αυτή την ωραία συζήτηση και την ωραία ατμόσφαιρα, κύριος Κάζ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η μικρομεσαίες είναι η κεντρία δύναμη τη Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Πρέπει λοιπόν να τις ενισχύσουμε και να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης στην Ένωση. Αυτό λοιπόν στα πλαίσια μια ελεύθερη αγοράς και ελεύθερη αγορά εννοώ μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένωσης. Πρέπει να δώσουμε στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν περισσότερες δυνατότητες, περισσότερα μέσα και να άρουμε τους φραγμούς και τα εμπόδια, ιδιαίτερα αυτά που απορρέουν από την χρηματοοικονομική κρίση. Όπως υπόθηκε νωρίτερα, για το ενωμένο Βασίλειο, όταν αποφασίσει μια χώρα να φύγει από την Ένωση, το φεύγω σημαίνει φεύγω. Όταν λοιπόν ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις είναι σημαντικό να κατανοήσουν ότι εκτός Ένωσης δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία, των οποίων απολαμβάνουν οι χώρες μέλη που είναι μέλη της, ε, της Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την επιχειρηματικότητα η οποία πρέπει να είναι τμήμα ακριβώς των κοινωνιών μας και γι' αυτό χρειαζόμαστε σωστές επιλογές. Η επιλογή για το επιχειρήν πρέπει να είναι ελκυστική. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα το πνεύμα κοινοτομία μας ε, γιατί έχουμε πολλέ προκλήσει να αντιμετωπίσουμε και δεν έχουμε κάνει ακόμα αρκετά. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι με την εμπειρία μας και την σκληρή μα δουλειά και εδώ να ευχαριστήσω του ηγητέ, νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο για τις μικρομεσαίες ιδιαίτερα σε χώρες και μέρη όπου κυριαρχεί η ανεργία και να λύσουμε το πρόβλημα ανεργίας που αντιμετωπίζει η Ένωση αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πάβελ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω τον συγητή για την συνεργασία που είχαμε στην προετοιμασία αυτής της έκθεσης. Και εγώ είμαι υπέρμαχος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γιατί πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε την ανάπτυξη οικονομική και κοινωνική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να στηρίξουμε και να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο και προϋποθέσεις ε, για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με καλύτερη πληροφόρηση, καλύτερη χρηματοδότηση και απλοποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε κλατικές προμήθειες και διαγωνισμούς. Να καταπολεμήσουμε την ε, διαφθορά, την απάτη και να δημιουργήσουμε ένα προβλέψιμο και σταθερό νομικό πλαίσιο. Αυτό ζητείται από πολλούς και στη χώρα μου, αλλά όχι μόνο. Πολλοί θα μου απαντήσουν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να προτείνει κανείς αυτά τα μέτρα από το να τα υλοποιήσει. Θεωρώ παρόλα αυτά ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει πραγματικά να υλοποιηθούν άμεσα αν θέλουμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για να υπάρχει δεμητός ανταγωνισμός και για να αυξηθούν οι δεξιότητες και τα προσόντα των εργαζόμενων στο εσωτερικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεισφέρουν και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αλλά και όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα κατάρτισης για να υπάρξει καλύτερη αντιστοιχία μεταξύ των αναγκών της αγοράς και της προσφοράς των προσόντων και των δεξιοτήτων σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μειώσουμε το κόστος και τις αμοιβέ των εργαζομένων γιατί αλλιώς θα δημιουργήσουμε περισσότερη επισφάλεια στην Ευρώπη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να έχουν ίσες αμοιβέ για άντρες και γυναίκες. Η Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει πολλά να κάνει για να στηρίξει ένα πλαίσιο αποτελεσματικό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να στηρίξει τις επενδύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Αντιπρόεδρε, ο εισηγητής μας παρουσιάζει ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλύπτουν το 90% της επιχειρηματικότητας ε, στην Ευρώπη και είναι στην πηγή ενός μεγάλου τμήματος της ανάπτυξης και της ε, καινοτομίας. Η έκθεση είναι εξαιρετικά σημαντική διότι προσφέρει ιδέες, προτάσεις και συμπεράσματα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης αναλύει και κάποιες ε, λιγότερο <clears throat> εύκολες ε, λύσεις όσον αφορά παραδείγματο χάρη την ε, αναδυστυχία μεταξύ των αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εργαζόμενων στην αγορά. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φανίου Χάιζεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, εισηγητές, καταρχάς θέλω να πω ότι συμφωνώ με τους είναι η ασμομηχανή μας σε όλα τα κράτη-μέλη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία τώρα που παίρνει μπρος η οικονομία να παίρνουν μπρος και οι εταιρείε και χρειάζονται χρηματοδότηση για το λόγο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται με την Ένωση Κεφαλαγορών και μας κάνει σημαντικές προτάσεις, δεν λέω, όντως θα συζητήσουμε και στη συνέχεια για ε, το ενημερωτικό δελτίο ε, την έκθεση του κυρίου Πέτερ Γέζε. Είναι μια καλή κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Μπορεί να βοηθήσει και ε, αυτό με τις κινητές αξίες για τα κεφάλαια κινδύνου κτλ. Όλα αυτά είναι σημαντικά στοιχεία, δεν αντιλέγω αλλά για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ε, δεν ε, τους βοηθάει πολύ. 80% είναι εξάρτησή τους ακόμα από τις τραπεζικές ε, δανειοδοτήσεις και επειδή είμαι και εισηγήτρια για ένα σχετικό θέμα, θέλω πάρα πολύ να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες, το crowdfunding, ε, οι πλατφόρμες επιγραμμικές για να δανείζονται οι πολύ μικρές επιχειρήσεις όπου έρχονται σε άμεση επαφή οι επενδυτές με τις εταιρείες και θα ήθελα ε, να δούμε και το FinTech ε, και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μήπως μπορεί να δοθεί ιδιαίτερη στήριξη για τη χρηματοδότηση αυτή. Και τέλος θέλω να συγχαρώ τους δύο συγητές για την καλή έκθεση τους. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λοπές Περμέχο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι μικρομεσαίες είναι σημαντικές στη διαθρώση του παραγωγικού μας μοντέλου, στην διατήρηση των θέσεων απασχόλησης και της παραγωγής. Παρ' όλα αυτά απειλούνται από τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Αφενός, οι τραπεζικές συγκεντρώσεις μετά από την διάσωση όπου παλαιότερα είχαμε ένα μοντέλο τράπεζας διαφοροποιημένο με μικρές τράπεζες, δημόσιες τράπεζες που χρηματοδοτούσαν τις μικρομεσαίες. Τώρα έχουμε μόνο μεγάλες τράπεζες οι οποίες είναι απομονωμένες από την πραγματική οικονομία που διοχετεύουν τις πιστώσεις στην κερδοσκοπία υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων και εις βάρος των μικρών. Και η έλλειψη ζήτησης που προκλήθηκε από τις περικοπές μείωσε τα εισοδήματα των μικρομεσαίων, οδηγώντας τες σε μια σοβαρή οικονομική κατάσταση. Η Ένωση λοιπόν Κεφάλαια Αγορών δεν αποτελεί την λύση θαύμα για αυτά τα προβλήματα όπως θέλει ο συγγητής. Αντίθετα, ρίχνει λάδι, λάδι στην φωτιά της ε, χρηματοδότησης, προκαλώντας μελλοντικέ ε, κρίσεις παρόμοιες με αυτές ε, οι οποίες τις πλήττουν τώρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ναι. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Απόψε άκουσα θετικές παρεμβάσεις από άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για την τύχη των μικρομεσαίων. Αυτό με ευχαριστεί. Βλέπω όμως ότι ακόμα και σήμερα δύσκολα ή με δυσκολία καταλαβαίνουμε τα πραγματικά προβλήματα των μικρομεσαίων στην Ευρώπη. Δεν είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και για άλλη μια φορά στο εσωτερικό της Ένωσης κοιτάμε το δάχτυλο και όχι τα πραγματικά αίτια, δηλαδή το χρηματοοικονομικό σύστημα και τις τράπεζες. Αυτό λοιπόν το νομικό πρόβλημα έχει ένα συγκεκριμένο όνομα, το ευρώ, το ενιαίο νόμισμα του ευρωπαϊκό, το οποίο βαραίνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μας το λέει η ίδια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα στις εκθέσεις της που αφορούν τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν ευκολύνονται στην πρόσβαση χρηματοδότησης, δεν ευκολύνονται για την έλλειψη πελατών, δεν ευκολύνονται στην, ε, στις εξόδους για τα προϊόντα του. Σήμερα το ευρώ προκαλεί μεγάλη στρέβλωση στον ανταγωνισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για άλλη μια φορά, δεν το λέω εγώ, το λέει το Νοτού και ο ΩΣΑ. Μας λένε κάτι το πολύ απλό, ότι σήμερα οι χώρες του Βορρά και οι μικρομεσαίες του Βορρά λειτουργούν με συναλλαγματική ισοτιμία υπερεκτιμημένη κατά 15-20%. Αντίθετα, για τις επιχειρήσεις του Νότου ισχύει το αντίστροφο. Αυτό είναι ε, ξεκάθαρο ότι με αυτή την ανισορροπία δεν υπάρχει μέλλον. Αυτέ οι ανισορροπίε θα διευρυνθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσει θα συνεχίσουν να κλείνουν. Εξάλλου και η λιτότητα που έχει επιβληθεί από την Ευρώπη στις ε, χώρες μέλη που έχει καταστρέψει τη ζήτηση και την κατανάλωση αλλά και τα εισοδήματα δεν βοήθησε καθόλου βέβαια τις μικρομεσαίες. Και αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα που σήμερα η Ευρώπη αρνείται να κοιτάξει. Εγώ λοιπόν δεν αποδέχομαι στο να συμμετάσχω σε αυτό το ολέθριο παιχνίδι. Και να σας πω το εξής, θα πρέπει να κάνουμε κάτι το πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το μοναδικό. Δηλαδή θα πρέπει να εξαρθρώσουμε, να καταστρέψουμε την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Μπέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση αυτή είναι μία από τις ατελείωτες εκθέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πέρα από τις δηλώσεις αρνούνται οι πολιτικοί μας να κάνουν κάτι για τον ανταγωνισμό, τον αθέμητο από μέρους της Κίνας. Βλέπουμε ότι στην Γαλλία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πλήττονται από την φιλελευθερισμό αλλά και από τον κρατισμό και από τη μία μεριά δεν δίνεται έμφαση στην πραγματική οικονομία, βαριά φορολογία, γραφειοκρατία και ανασφάλεια νομική, κάτι που είναι απαράδεκτο και πάρα πολύ δύσκολο να το αντέξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν έχουν πρόσβαση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις κρατικές προμήθειες και θα πρέπει πραγματικά να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και όχι τις τράπεζες. Σήμερα 22% είναι η φορολογία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ μόνο 8% για τους μεγάλους ομίλους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πίπερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε θα μπορούσαν να είναι τόσο ωραία. Καλές εκθέσεις για το μέλλον ε, των μικρομεσαίων, χρηματοδότηση, θέσεις απασχόλησης στο ε, κέντρο της προσοχής. Ευχαριστώ τους δύο εισηγητές Κάρας και Κρασνοντεύσκη που πραγματικά ασχολήθηκαν ε, τόσο ελπιδοφόρα με το θέμα. Θα μπορούσαν να είναι τόσο ωραία αν δεν βλέπαμε και άλλα μηνύματα αυτή την εβδομάδα. Αριστεροί, πράσινοι και φιλελεύθεροι θέλουν ε, μια νέα εκδοχή της ε, οδηγίας για την προστασία της μητρότητας αυτό είναι ένα θέμα εθνικό και επιβαρύνει ιδιαίτερα τι μικρομεσαίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ρυθμίσει τα των γονέων και να συμμετέχουν και οι, πατέρες αυτή την υπόθεση, να φροντίζουμε του ηλικιωμένου μας. Αλλού ζητούμε κατώτατου μισθού αυτή τη βδομάδα, θέλουμε μια, ε, ε, ε, ασφάλεια για την ανεργία πανευρωπαϊκή και ε, θεωρούμε διαβολικό και σατανικό κατασκεύασμα το outsourcing, την εξωτερική ε, ανάθεση. Ε, δεν μας αφύπνισε το Brexit, ήταν πραγματικά αφυπνιστικό, αλλά εμείς τι κάνουμε, σκάβουμε το λάκκο μας. Ε, παραβιάζουμε την επικορικότητα, επιβαρύνουμε τις επιχειρήσεις. Δυστυχώς και αυτός είναι ο απολογισμός της εβδομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό θα πρέπει όσοι ασχολούνται με τις μικρομεσαίες ε, ε, να ανοίξουν τα χαρτιά τους όπως εμείς σήμερα και να τα πούμε με το όνομά τους. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δύο λεπτά. Φερνάντε, Καλησπέρα σας. Τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω να ευχαριστήσω τους ηγητές και να χαιρετήσω ε, τον κύριο Ντομπρόφσκης για την παρουσία του. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συζήτηση αυτή και θα πρέπει να προλιάρουμε τώρα το έδαφο έτσι ώστε η πραγματική οικονομία στην Ευρώπη να ανακάμψει, να βελτιώσει την απασχόληση και την ευημερία τελικά όλων των Ευρωπαίων. Είναι γεγονό ότι υπάρχουν πολύ μικρέ προκλήσει που πρέπει και να τι αντιμετωπίσουμε, να αναθεωρήσουμε όλε τι κλαδικέ πολιτικέ που προωθεί η Κομισιόν, τηλεπικοινωνίε, ενέργεια για να βελτιωθούν οι προοπτικές ανάπτυξη. Αλλά και οι μακροοικονομικές πολιτικέ χρειάζονται αναθεώρηση, όχι μόνο νομισματική και άλλε η Ένωση Κεφάλαιο Αγορών για να διευκολύνει τη χρηματοδότηση και βεβαίως φορολογική πολιτική. Διότι μέγα τμήμα των προβλημάτων τους είναι ότι δεν υπάρχει ζήτηση. Άρα και τα δημοσιονομικά πρέπει να λυθούν. Και όλα αυτά βελτιώνοντας ε, την δυνατότητα ανταγωνισμού για να μην υπάρχει φορολογικό dumping από τις μεγάλες επιχειρήσεις που μας απασχόλησαν προηγουμένως. Η έκθεση είναι στη σωστή κατεύθυνση, μπορεί να βοηθήσει τη Γομισιόν και τα άλλα θεσμικά όργανα να συνεργαστούν και να συνεχίσουν και η ομάδα μου και εγώ προσωπικά θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ εύστοχη και επίκαιρη η έκθεση. Επιτρέψτε μου μερικά δευτερόλεπτα να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Επίτροπο που τον φέραμε εδώ 11 η ώρα να ακούει ε, το UKIP και ε, το εθνικό μέτωπο που είναι ντροπή και έσχος και για το Κοινοβούλιο και για όλους τους Ευρωπαίους. Εμείς εδώ δουλεύουμε ώρες ολόκληρες χρόνια τελείωτα και είναι αφόρητο να ακούμε τέτοια πράγματα μίσους που δηλητηριάζουν τους πολίτες που εκπροσωπούν το χειρότερο έσχος στην Ευρώπη και είναι πραγματικά ντροπή και ε, θα ντρεπόταν ο Ντεγκόλ, ο Τσόρτσιλ και οι πατέρες της Ευρώπης. Έχει φτάσει σε ένα τελείως αφόρητο και ανυπόφορο επίπεδο πια αυτή η ιστορία. Αυτά τα λίγα και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φερνάντες, λέει πρόεδρος. Ένα μενόμενο ήτανε. Αν ε, χρησιμοποιείτε το χρόνο σας για να απευθύνεστε σε άλλους ευρωβουλευτές, σηκώνονται μπλε κάρτες. Τώρα θέλετε να απαντήσετε σε μια ερώτηση από μπλε κάρτα. Μάλιστα. Thank you, madam. Thank you, uh, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Φερνάντε. Είπατε κάτι για το UKIP. Ανόητο μου φάνηκε. Ο, ο επίτροπο κάθε εδώ αργά, είπατε. Μεγάλο μισθό έχει, οπότε δεν είναι κακό να ακούσει και Εμά τους λαϊκιστές και τα λοιπά, ξέρω δεν φορολογείται και τόσο. Είναι καλύτερο να είναι κανείς ε, ε, από εσά που είστε μη λαϊκιστή. Ευχαριστώ. Δεν είδα κάποια ερώτηση εδώ. Κατανοείτε ότι, κοιτάξτε, μπλε σημαίνει ερώτηση, έτσι, ώστε να λάβετε κάποια απάντηση ενδεχομένω. Αλλά τέλο πάντων, θέλω να ακούσω την απάντησή σα. Ναι, βεβαίω θα είμαστε όση ώρα χρειάζεται εδώ. Γιατί αυτό το εγχείρημα, το εγχείρημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το καταστρέψετε εσεί, ούτε εσεί ούτε κανένα άλλο σαν και εσά. Όλοι οι πολίτε είμαστε εδώ και στηρίζουμε από την Αστούρια, στην περιοχή μου, την ε, Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κυριαρχία. Περιού ο λόγο. Εσεί αυτό προσπαθήστε εδώ να το καταστρέψετε. Και το κυριότερο είναι ότι καταστρέφετε και εσεί σα τι χώρε. Πολύ ωραία, λέει η Πρόεδρος. Λοιπόν, Ελπίζω να μιλήσει για το θέμα ο επόμενο ομιλητή μα, ο κ. Σιλικιώτη. Παρακαλώ. Στην έκθεση για αξιοποίηση του δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων συνεργασία, το Κοινοβούλιο επικαλείται και πάλι την ελεύθερη αγορά ω φάρμακο δια πάσα νόσου. Επικεντρώνεται στη μείωση του λεγόμενου κόστου εργασία για πρόθεση νέων θέσεων εργασία στι μικρομεσαίε επιχειρήσει και σε ευελιξία στην αγορά εργασία δεν παραβλέπουμε τι καλέ προθέσει των εισηγητών και τι βελτιώσει που έγιναν στο κείμενο. Η αναφορά στη διασφάλιση τη προστασία των εργαζομένων, σε οποιαδήποτε αύξηση τη ευελιξία και η στήριξη τη ανάπτυξη εταιριστικών επιχειρήσεων μα βρίσκουν σύμφωνο. Διαφωνούμε όμω με την γενική φιλοσοφία τη έκθεση. Το γενικό πλαίσιο που προτείνεται για να αξιοποιηθούν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει για δημιουργία θέσεων εργασία δεν διασφαλίζει τη δημιουργία νέων αξιοπρεπών και μόνιμων θέσεων ούτε γίνεται λόγος για συλλογικά εργασιακά δικαιώματα δηλαδή την κοινωνική ασφάλιση τη συλλογική διαπραγμάτευση και τις συλλογικές συμβάσεις το φάρμακο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας και της απορρίθμισης εργασίας για δίθεν οικονομική ανάπτυξη απότυχε παταγωδώς αφού τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην ένωση. Σας ε, τώρα το λόγο έχει η κυρία Φων Στόρχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άρα σήμερα μιλάμε για τη χρηματοδότηση, λέει, μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με ορισμένα από την έκθεση. Βεβαίω είναι η ραχοκόκυλια τη κοινωνία. Οι μικρομεσαίε δημιουργούν τι περισσότερε θέσει εργασία, υφίστανται το μεγαλύτερο βάρο από τη γραφειοκρατία και έχουν και προβλήματα χρηματοδότηση. Όλα αυτά ισχύουν. Και επίση όλοι υποφέρουν και από το ευρώ που είναι αυτός ο στενός κορσές, αυτός ο ζουλομανδίας, ε, όπως ε, είπε και ο κύριος Τζάνι, ε, υποφέρουμε από αυτό το νόμισμα, εν πάση περιπτώσει. Οι προτάσεις στην έκθεση για τη βελτίωση της κατάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν με βρίσκουν σύμφωνοι. Οι μικρομεσαίες δεν χρειάζονται να τσουβάλει τώρα νέους κανονισμούς και ρυθμίσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αντίθετο χρειάζονται, λιγότερες ρυθμίσεις, ιδιαίτερα λιγότερες ρυθμίσεις από τις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει ε, ε, στραγγίσει τις χρηματαγορές από τις πολλές ρυθμίσεις και τα δισεκατομμύρια. Έχουμε παντού γραφειοκρατία στις χρηματαγορές και τράπεζες ζόμπι. Ε, αυτά είναι τα δηλητήρια ε, και οι αναθυμιάσεις της κρίσης του ευρώ και ε, ερχόμαστε να τα βάλουμε και στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων. Σταματήστε να σώσετε τις τράπεζες. Πάλι επιτρέψατε στην Ιταλία να σωθούν και στην Πορτογαλία. Τι θα γίνει τώρα αυτές οι τράπεζες ζόμπι, ε, να τις βγάλουμε από αυτόν τον ορό που τις έχουμε και τις γόνα σταγόνα σταγόνα, να σωθούν οι άνθρωποι, να σωθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιτέλους και να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σάλμπα. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπο, κύριε Επίτροπε, επιτρέψτε μου καταρχάς να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεσή του υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε όλη του τη διαδρομή ο κάρα ε, Κάρας υποστηρίζει αυτές τις επιχειρήσεις. όπως είπε και ο κύριος Δομπρόσκη και οι άλλοι συνάδελφοι είναι η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξής μας και της δημιουργία θέσεων εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό οποιαδήποτε έκθεση, οποιαδήποτε βοήθεια, οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να διευκολύνουμε την καθημερινή δουλειά των επιχειρήσεων αυτών, για να βοηθήσουμε την ανάπτυξή τους, είναι λίγο. Και αναμφίβολα ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες στην Ευρώπη και κυρίως στις χώρες του Νότου της Ένωσης είναι ακριβώς η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ή, καλύτερα, να το πω, τα διαφορετικά κόστη χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις στο σύνολο της Ευρωζώνης. Και αυτό είναι άδικο, γιατί κατά κάποιο τρόπο επηρεάζει και την παραγωγικότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σωστό να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω την Ένωση Κεφάλαια Αγορών Και νομίζω ότι αναμφίβολα οτιδήποτε αποτελεί διευκόλυνση στη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες θα είναι κάτι το οποίο αναμφιβόλως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σοβαρά και που απορρέει από την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκεί Πρόεδρος. Ο κύριος ε, Τσεντήλε έχει το λόγο. Παρακαλώ. Η κυρία Τσεντήλε. Πρόεδρε ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αναμφίβολα το σύστημα μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί το κυριότερο μοχλό ανάπτυξης. Ανάπτυξης που μας επιτρέπει να πετύχουμε τον κυριότερο στόχο, δηλαδή την πρόθεση της εργασίας. Είναι κεντρική λοιπόν σημασία η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Απλουστεύση, καινοτομία, μεγαλύτερη διάθεση κονδυλίων, καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ, μαύρη οικονομία Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη και συνεχόμενη κατάρτιση για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει να ανοίξουμε νέες δεξιότητες, επαγγελματικές, ανάλογα με τη ζήτηση που υπάρχει για να κερδίσουμε νέο περιθώριο αγορών. Πρέπει να έχουμε και δίκαιες ε, φορολογικές πολιτικές, αντικυκλικές πολιτικές, πολιτικές με στόχο την ανάπτυξη, για να προωθήσουμε εργαλεία τα οποία θα μπορέσουν να είναι αποτελεσματικά όσον αφορά την ένταξη στην αγορά εργασία των πιο αδυνάμων. Και τέλος, χρειάζεται περισσότερη κοινωνική ευθύνη. Διακόπτη Πρόεδρος, για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς τις ε, μορφές εργασίας της ε, προβληματικέ. Σας ευχαριστώ. Για ένα μισό λεπτό ζητώ συγγνώμη μην χρησιμοποιείτε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο κάρα, και όλου όσου συνεργάστηκαν για αυτή την εξαιρετική έκθεση. Χαιρετίζω επίση και τον την πρόθεση του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επέκταση του Ταμείου και των επενδύσεων που ήδη έχει χρηματοδοτήσει και στηρίξει 200.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στηρίζω επίσης τις προτάσεις της έκθεσης αυτής που αφορούν την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης που προσφέρει η εσωτερική αγορά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι ο αντιπρόεδρος πρόφτης είπε κάτι που είναι ουσιαστικό. Χρειαζόμαστε περισσότερο παρά ποτέ την ένωση των κεφαλαγορών. Σήμερα, εν ώψη του Brexit, αυτό γίνεται επίγον. Και ακριβώς επειδή η ψηφιακή οικονομία επεκτείνεται, θα πρέπει να υποβάλουμε νέες προτάσεις που να στοχεύουν τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να στηρίξουμε την καινοτομία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σήμερα στην Ευρώπη εργάζονται με συγκεκριμένες εφαρμογές της ψηφιακής οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την τήρησατε και τον χρόνο σας. Ένα λεπτό, τον κύριο Ζαμανάτο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σημαίνει στήριξη της απασχόλησης, ιδιαίτερα απασχόληση των νέων και υποστήριξη κοινωνική συνοχή. Γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να επικεντρωθούμε στι μικρο, μικρομεσαίες, στις μακροεπιχειρήσει και στις startup, διευκολύνοντας ακριβώ την κατάρτιση και την εξειδίκευση. Το πρόγραμμα Εράσμους για του νέου επιχειρηματίε που του βοηθάει στις γνώσεις και στις απαραίτητες δεξιότητες για να ξεκινήσουν και να δικήσουν μια επιχειρήση θα πρέπει περαιτέρω να αναπτυχθεί και να κοινοποιηθεί, να διαφημιστεί. Θα πρέπει επίσης να βοηθήσουμε και τους πιο αδύναμους να δημιουργήσουν μικρομεσαίες. Η συμμετοχή, ας πούμε, των μεταναστών στον ε, κόσμο της εργασίας είναι μια μεγάλη ανάγκη. Αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο υποχρησιμοποιείται ακόμα λόγω της ε, δυσκολίας ε, λήψης ε, άδειας εργασίας, λόγω των διακρίσεων και λόγω των γραφειοκρατικών φορολογικών επιβαρύσεων και της δυσκολίας στην πρόσβαση στην χρηματοδότηση και έλλειψης ακριβώς σταθερότητας στην διαμονή. Ευχαριστώ πολύ. Για 1,5 λεπτό δίνω το λόγο στην κυρία Τόμιτς. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Κάθε φορά που αναφερόμαστε στο θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φτάνουμε στα ίδια προβλήματα και δυσκολίες. Το θέμα της χρηματοδότησης. Θα ήθελα να προσθέσω όμως και κάτι άλλο σε αυτά που ακούστηκαν. Η χρήση μέσων από ευρωπαϊκά προγράμματα θα ήταν επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν ίσως και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς, σε υποβολή προσφορών για κρατικές προμήθειες και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να απλοποιήσουμε και τις διαδικασίες έτσι ώστε να μειωθεί το γραφειοκρατικό τους βάρος. Χρειαζόμαστε επίσης και θύλακες, πλατφόρμες, τις οποίες να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ελαχιστοποιήσουν το κόστος τους ε, θέτοντας από κοινού μέσα και προσωπικό. Έχω πολλές προτάσεις να κάνω. Χρειαζόμαστε ένα καλύτερο περιβάλλον με περισσότερη ευελιξία για να μπορέσουν ε, να δραστηριοποιηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει επίσης να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Πάνοβα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε εδώ για τους επιχειρηματίες, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης χρειάζεται χρηματοδότηση και ίσες ευκαιρίες για να αναπτύξουν τις ιδέες τους στην δική μας ευρωπαϊκή αγορά. Δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο σε μία πηγή χρηματοδότησης. Θα πρέπει να υπάρχει κρενοτομία, δημιουργικότητα, ευελιξία, όπως είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σήμερα και δεν υπάρχει μία λύση που να ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες. Χρειάζονται λύσεις και προσαρμογές της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που να μπορεί να ανταποκριθεί στις δικές τους ανάγκες. Και βεβαίως αυτές οι προτάσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Χρειαζόμαστε ταχύτατη προσαρμογή στην πραγματικότητα και δράση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ανάπτυξη την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων αποσχόλησης. Πρέπει να στηρίξουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης, ε, τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω των κεφαλαγορών και να δημιουργήσουμε νέες πρωτοβουλίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν είναι δυνατόν να αρκεστούμε στις σημερινές λύσεις. Χρειαζόμαστε νέες καινοτόμες λύσεις και μπορούμε να τις παρέχουμε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον τελευταίο μιλητή για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Κάρας, πολύ καλή έκθεση του για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ κύριε Ντομπρόμψκης για την παρουσία σας και για την προσωπική σας στράτευση σε αυτή την υπόθεση. Όταν μιλούμε για την Ένωση Κέφαλε Αγορών υπάρχουν διάφορα μέσα και εργαλεία που έχουμε στην εργαλειοθήκη μας, αλλά θα πρέπει να τα αξιοποιούμε όλα. Διότι είδαμε και από τη χρηματοπιστωτική ε, κρίση ότι δυσκολεύονται να χρηματοδοτηθούν οι μικρομεσαίες. Το ακούσαμε από όλους τους ομιλητές ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα. Ακούσαμε σήμερα ότι ο κύριος Γιούνκερ ε, θέλει να αυξήσει τη χρηματοδότηση του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Πολύ ωραίο αυτό και για τις μικρομεσαίες και για εκείνους που πήραν χρήματα από την πρώτη δόση. Σήμερα άκουσα επίσης και για την υλοποίηση ε, των κανόνων της Βασιλείας. Ε, δεν διευκόλυνε αυτό τις μικρομεσαίες να χρηματοδοτούνται. Ε, μιλώ για τις πραγματικές ανάγκες για κεφάλαια κίνησης και ρευστότητα. Και τώρα ε, υπάρχει και η τέταρτη οδηγία για τις κεφαλικές ε, απαιτήσεις που έρχεται να ε, κάνει πιο σκληρά τα κριτήρια της Επιτροπής της Βασιλείας. Αν συγκρίνουμε τις ευρωπαϊκές εταιρείε με τις αμερικανικές θα δείτε ότι οι Αμερικανοί έχουν πολύ λιγότερες υποχρεώσεις. Και εμείς τους αλλάζουμε τα φώτα μέχρι να τις χρηματοδοτήσουμε. Πρέπει να βρεθεί κάποια λύση, εν περιπτώσει να το έχετε υπόψη σας αυτό κύριε Ντομπρόφσκης. Ε, η Πρόεδρος, πάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Μαριάς, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 99,8% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργούν το 55% του συνολικού ΑΕΠ της Ένωσης και απασχολούν 75 εκατομμύρια πολίτε συμβάλλοντα έτσι στην οικονομική κοινωνική και περιφερειακή συνοχή. βέβαια σε χώρε όπω η ελλάδα ο τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει πληγεί ιδιαίτερα από τι δυσμενεί επιπτώσει του μνημονίου ενώ μέχρι το 2015 εξαφανίστηκαν 244.000 σαράντα και οδηγήθηκαν στην ανεργία 842.000 άτομα παράλληλα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν περιορισμένη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό ενώ η στήριξη που αναμένεται να δοθεί από το ευρωπαϊκό ταμείο στρατηγικών επενδύσεων για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν φαίνεται ότι μπορεί να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. προκειμένου όμως να αρθεί κάθε εμπόδιο στην ανάπτυξη και στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων θα πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν τα προγράμματα του ευρωπαϊκού ταμείου στρατηγικών επενδύσεων ενώ οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες. ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βιέγας, επόμενος ομιλητής. Ε, εμείς δεν αμφισβητούμε την ανάγκη Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τι μικρομεσαίε. Αυτό είναι σημείο κλειδί. Όμως δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα χωρίς τη σωστή διάγνωση. Δηλαδή θα πρέπει να ξεκινήσουμε την προσπάθεια επίλυσης αυτού του προβλήματος λαμβάνοντα υπόψη την κατάσταση των τραπεζών. Το κάνουμε όμω αυτό χωρί να λάβουμε κανένα αντίδραγμα από την κατάσταση που έχουμε μέχρι τώρα. Και η κατάσταση στην αγορά κεφαλαίων ε, δείχνει ότι έχουμε όλο και περισσότερο επιχειρήσει που είναι όλο και πιο δύσκολο να αποτύχουν να πτωχεύσουν. Πρέπει να πούμε ότι τα τραπεζικά συστήματα είναι κυρίως εθνικά με περιφερειακές βάσεις. Γι' αυτό ακριβώ χρειαζόμαστε την ύπαρξη άλλων τραπεζών όπω τράπεζα για τη βοήθεια τη ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Φτάσαμε στο τέλος της διαδικασίας Κατσιά και τώρα θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο του Πρόσκης. Κυρία Πρόεδρε, ξέρετε μέλη του Κοινοβουλίου. Μετά από αυτήν την ανταλλαγή απόψεων είμαι πεπισμένος ακόμα περισσότερο ότι πρέπει πραγματικά να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Άμεσες πρωτοβουλίες για ενίσχυση του τρόπου των επενδύσεων είναι κάτι που θα αποφέρει άμεσα αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικές οι προτάσεις που κάνουμε σήμερα και βεβαίως οι νέες προτάσεις τις οποίες θα συμφωνήσουμε για πιο φιλόδοξη δράση που βασίζονται στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έγινε αυτή η συζήτηση όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τους τρόπους να στηρίξουμε τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Συζητήσαμε πολύ σημαντικά θέματα και υποβάλλατε πολύ σημαντικές συστάσεις. Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει όλες αυτές τις προτάσεις για αυτόν τον τόσο σημαντικό τομέα. Τώρα θα δώσω το λόγο στους εισηγητές προς τον κύριο Καρά. Κύριε Καράς, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε και κύριοι. Τι μας έδειξε η συζήτηση. Και ο αριθμός των ομιλητών τέτοια ώρα μάλιστα. Τι μας έδειξε. Ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ενίσχυση χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πόσο σημαντική είναι για μας. Δεν χρειάζεται να τονίσω τι σημαίνει για την εσωτερική αγορά, για την ανάπτυξη της οικονομίας και της απασχόλησης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σήμερα στη συζήτηση, τους και που συμμετείχαν στην εκπόνηση της έκθεσης και την ε, πλαισίωσαν καθόλου την κατάρτισή της. Θα ήθελα όμως να πω και αυτό. Η απόψινή συζήτηση επικεντρώθηκε στη χρηματοδότηση και τη διαφοροποίηση των πηγών των μικρομεσαίων στην Ένωση Κεφαλαιογορών. Αυτό είναι το θέμα μας. Και όχι γενικός και ορίστος. Η Ένωση Κεφαλαίου Αγορών θα πρέπει να διαμορφωθεί έτσι και να την αντιλαμβανόμαστε ως ένωση χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. Και θα πρέπει η ροή των κεφαλαίων και των δανείων προς τις μικρομεσαίες όχι απλώς να απλοποιηθεί αλλά και να διευρυνθεί. Και γι' αυτό φυσικά είναι αυτονόητο να διευρυνθεί το ΕΦΣΥ, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Και μέχρι τώρα η θηρίδα για τις μικρομεσαίες ήταν σημαντική. Εδώ ανήκει και το πρόγραμμα Εράσμος για ε, μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Εδώ ανήκει επίσης η υλοποίηση του Small Business Act ή το Single Market Act, όλα αυτά τα νομοθετήματα για την εσωτερική αγορά. Και εδώ ανήκει και ε, μία εφαρμογή των κριτηρίων της Βασιλείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό που ισχύει στις Ηνωμένε Πολιτείε και στην Ευρώπη. Όπου 80% της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων ε, είναι από τις τράπεζες. Δεν λέω ότι είναι τέλεια η έκθεση ολοκληρωμένη, αλλά είναι σημαντικό βήμα προς την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών, που να την αντιλαμβανόμαστε ως Ένωση Χρηματοδότησης, επαναλαμβάνω, της πραγματικής οικονομίας. Δεύτερο συγητής, ο κύριος Κράσνοτεύσκη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για όλα τα πολύτιμα σχόλια που άκουσα κατά διάρκεια της συζήτησης. Να προσθέσω κάτι άλλο. Είπαμε πολλά για την χρηματοδότηση, για την πρόσβαση στην χρηματοδότηση και πόσο σημαντική είναι για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων αυτών επιχειρήσεων. Να πω στο το εξής επιπλέον κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε μέχρι τώρα εδώ στη συζήτηση. Νομίζω ότι όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν, δεν θα πετύχουμε δηλαδή την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων χωρίς να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα. Πρόσφατα είχαμε μια έρευνα μεταξύ των φοιτητών στη Γερμανία που τους ρωτούσε αν θα τους ενδιέφερε να είναι αυτοαπασχολούμενοι και νέοι επιχειρηματίες. Οι γυναίκες φοιτητέ, η πλειονότητά τους είπαν ότι ήθελαν να δουλέψουν για το δημόσιο. Το ίδιο και οι άντρες. Αυτή ήταν η πρώτη επιλογή και των δύο. Δεύτερη επιλογή μεταξύ των γυναικών ήταν τα πολιτιστικά ιδρύματα και οι γυναίκες και οι άντρες ε, ως δεύτερη επιλογή επέλεξαν την αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό μας δείχνει ότι το πνεύμα επιχειρηματικότητας θα πρέπει να προωθηθεί στην Ευρώπη. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν αποτελεί προτεραιότητα. Επειδή ο κόσμος θεωρεί ότι οι καλύτερες σταδιοδρομίες, οι καλύτερες ευκαιρίες ε, βρίσκονται ακριβώς στο δημόσιο, στις θέσεις εργασίας που προσφέρει το δημόσιο. Αυτό είναι ένα πρώτο σχόλιο. Ένα δεύτερο σχόλιο είναι κάτι το οποίο ανέφερα προηγουμένως, αλλά θα ήθελα να επανέλθω. Στην έκθεσή μας λέμε ότι Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων από χώρα σε χώρα και υπάρχουν και διαφορετικοί φραγμοί που αντιμετωπίζουν αυτού του είδους επιχειρήσεις. Και το είδος εμποδίων είναι και αυτό διαφορετικό. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτές τις διαφορές, γιατί τα προβλήματα είναι διαφορετικά ανάλογα με το αν βρίσκεται μια επιχείρηση στην Πολωνία ή στον Μπάντεν Βίρτεμπεργκ. Και αυτό η στον μπαντεν βιρτεμπερκ και αυτο η κομισιον θα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη της. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λεκή Πρόεδρος, για αυτές τις ιδέες σας. Κύριοι βουλευτές, τώρα θα κλείσω την συζήτηση.